Ladies and gentlemen, good morning. Καλημέρα σας. We would like to start now. Θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ο κύριος Λουίς Τεγκράντες ζητάει το λόγο όμως. Ορίστε. Εκτός μικροφώνου δεν τον ακούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα προκαταρκτικό ζήτημα αλλά σημαντικό η Επιτροπή μας που ασχολείται με τα εξωτερικά θέματα δεν θα μπορούσε και το λέω πρόεδρος ε, ε, της Αντιπροσωπής για τις σχέσεις με τις ε, χώρες της Ελληνικής Αμερικής τη συμπαράστασή μας για το σεισμό στο Εκουαδόρ που άφησε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, τρομερή τραγωδία με φοβερές ανθρώπινες και ηλικές απώλειες και ζημιές. Είχαμε ε, μια πολυμερή συμφωνία όπως και με την Κολομβία και το Περού και με το Εκουαδόρ και θα ήθελα να εκφράσω αυτή την συλλογική μας συμπαράσταση. Ε, θα έλεγα είτε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή και να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και τη συμπαράστασή μας στον λαό του Εκουαδόρ που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται πολύ σκληρά. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, λέει ο Πρόεδρος, ότι εκφράζουμε αλληλεγγύη και συμπόνια με τον κόσμο εκεί, με τις οικογένειες που θρυνήσαν θύματα, πολλά θύματα. Και φαίνεται ότι αυξάνεται ο ρυθμός ε, των ε, νεκρών. Και βλέπουμε φυσικά παντού πως ε, η μητέρα φύση είναι παντοδύναμη σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους και πώς είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες δραματικές καταστάσεις. που φαίνεται ότι είναι αδύνατες ε, παρά το γεγονός ότι και στην Ιταλία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπήρξαν τέτοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία. Να σηκωθούμε λοιπόν όρθιοι για μια στιγμή να τιμήσουμε τα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 Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία στο σημείο αυτό για τις Φιλιππίνες. Τρεις ψηφοφορίες έχουμε να κάνουμε. Το θέμα της συνένεσης. Εδώ ο εισηγητής δεν έχει κάτι να μας ε, ανακοινώσει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 52 η ψηφη υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία τώρα. συμπεράσματα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο για τη συνεργασία για να λεφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Κροατία, λοιπόν, ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας. Πέντε δύο ψήφοι υπέρ, δύο α, ψήφοι κατά, έξι αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πέντε στην έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και εισηγητές. Νομίζω ότι επιχειρήσαμε να συνενώσουμε και να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση που δείξατε, για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε κάθε ε, μικρό στοιχείο και επιμέρους στοιχείο. Νομίζω όμως ότι το πνεύμα και το περιεχόμενο ε, περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις. Δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε και με υπερβολικό επίπεδο λεπτομέρεια στην έκθεση. Ας ψηφίσουμε. Υπάρχει πρόβλημα με την Ισπανική διερμηνία, με την Ισπανική διερμηνία δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά το θέμα των Φιλιππίνων. Εντάξει, πολύ ωραία. Μάλιστα. Διορθώθηκε το πρόβλημα. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά.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 κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία. Η 68 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Να... Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Χατζηγεωργίου. 14 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. αποχέ, απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ξανά 19 παρακαλώ υπέρ.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3... Πάρα πολλές υγραπλογές βουτικόφερ. 30 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 30. Να τις ψηφίσουμε όλες τις μπουτικόφερ λοχπίλερ ε, με μιας. Unblock. Να ψηφίσουμε την 21 μέχρι και την 33 παρακαλώ μαζί. Την 30, την 30, ναι. Γιατί την έχουμε ψηφίσει την 29. Να βάλουμε και τη Χατζηγεωργίου. 30 έως 36, υπέρ. Όχι. την 29-31, ε, αλλά τις υπόλοιπες έχουμε διαφορετικό. Εντάξει, ναι, την έχουμε ψηφίσει την 29, άρα 30 μέχρι 31. Με σας ρώτησα, συμφωνείτε, τέλος πάντων, να το ψηφίσουμε μία-μία, να ξεμπερδεύουμε. 30 υπέρ, κατά. Έλεγχος παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 35. Πέρας. Απορρίπτεται 28 υπέρ, 36 κατά. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η αποτέλεσμα. 1, 2, 3. Ταυτόσιμες. Πώς το εσύ γιατί είσαι αυτό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 5, 6, 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου. Έναρξη της ψηφοφορίας. Can I have these identical amendments? How is that possible? Yeah, nevertheless. The vote is closed. I would like to... Πέρας. It's uh, adopted by... Εγκρίνεται 57 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Äh, Και τώρα περνάμε στην έκθεση Να ξεκινήσουμε καταρχάς με την έκθεση Van Orden πρώτα. Το ζήτησε ο κ. Στοβιέσκη. Και δέχεται και ο κ. Van Orden. Κύριε Σιγητά, σχόλια έχετε να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε πολύ καλές συναντήσεις με τους συζητητές πολύ καλή συμφωνία μέχρι την δεκάτη ώρα που όλα άρχισαν να χάνονται κάπως, θα τα ξανασημαζέψαμε. Ελπίζω οι συνάδελφοι να ακολουθήσουν τη σύστασή μου για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Σμπροκ. ΔΕΒΕ 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. πέντε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. έξι, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87. 85 διορθώνει ο πρόεδρος. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. The vote is closed. 29 ψήφι υπέρ, 35 κατά. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. σύμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 100, 102 μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 107 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 108 υπέρ κατά άποχες 108 πάλι υπέρ κατά εγκρίνεται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 Άποχες. εγκρινετά. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρινετά. 114. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Άποχε. Έγκρινεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Άποχε, Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. απόχε. Εγκρίνεται. Η 13 η συμβαστική υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Πέρασα. 39 υπέρ, 27 κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον ε, κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Mm. Ναι, Μάσιμο, μου χρωστάς μια κράπα. Γι' αυτό. Πέρας. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ τώρα σου χρωστάω γράπα. Εγώ θα σε κεράσω. Στην υγειά σου θα πιάω.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 The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 58. 58 με 6 και δύο αποχές. Εγκρινούνται και συγχαρητήρια. Νομίζω ότι είναι η πρώτη έκθεση όπου νομίζω ότι έχουν περισσότερες τροπολογίες και αιτιολογικές σκέψεις ε, και αιτιολογικές σκέψεις και αιτιολογικές αναφορές από ό,τι για την ίδια την έκθεση. Ο κ. Κουζου. Ευχαριστώ. Η GUNGL έχει καταθέσει μια έκθεση μειοψηφία. Την έχουμε αποστείλει στη γραμματεία. Απλώς ενημερωτικά ήθελα να σας το πω. Ευχαριστώ πολύ. He Κατέφτασε. Α, να, εκεί είσαστε. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Οι διαστημικές δυνατότητες όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Έχετε κάτι να πείτε? Όχι, να ξεκινήσουμε αμέσως τις ψηφοφορίες. Συμβαστική 1, ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές γίνεται 2. Σημαστική 2 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σημαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Compromise 6. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές ε, δεν παίζουνε, δεν μας παίζουνε. Μα τι ψηφίσατε. Υπέρ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. 135 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Abstimmung Πέρας 32 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. 136 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 149 Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος ήταν 149. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 36 υπέρ, 29 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. κατά 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε εφόσον το επιθυμείτε. Πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 21 ψήφι κατά. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές. 170 παρακαλώ πάλι υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 190 Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. και 18 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. Πέρα. 23 υπέρ, 38 κατά. Απορρίπτεται. Αλλά ήθελα να είμαι σίγουρο. Ε. Κύριε Κασταλντό, 198 υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. Πέρας ψηφορίας. 39 υπέρ, 26 κατά. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Τριάντα μία υπέρ, 35 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να φέρουμε ένα καφέ στους σοσιαλιστές, μήπως. Και μία κρέπα. 32, που είχαμε μείνει στην 32, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 42 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45, 54 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ κατά άποχες έλεγχος για την 1. 24 υπέρ, 42 κατά απορρίπτεται. Οι 2 και οι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρασε. Με 29 υπέρ, 38 κατά, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν τώρα. Ist geschlossen. Πέρασε. 42 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, 10 αποχές. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ε, καταθέσει έκθεση μια ψηφία για το θέμα αυτό από την ομάδα της GUNGL. Τη στείλαμε στη γραμματεία. Πολύ σας ευχαριστούμε. Έχετε το δικαίωμα. Και περνάμε τώρα στην έκθεση Κόβατσεφ για τα Ηνωμένα Έθνη. Για τη Γενική Συνέλευση ο εισηγητής δεν θέλει να πάρει το λόγο, να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε τα 36 υπέρ. Α, έχω εγώ. Ποιος, ποιος μίλησε, ποιος, ποια. Μία πληροφορία. Έχω αποσύρει το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 190. Απλώς ε, αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω. 36. Ευχαριστώ. 36 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 190. Μόνο το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 91 υπέρ. Η 87 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος για την 87. Πέρας. 44 υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτός μικροφώνου. Κάποιο θέμα με την οθόνη. Ready. Kompromiss <laughs> eh? 9, υπέρ. Ή 100 λοιπόν. Τραπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά ας το ελέγξουμε. Πέρας. 41 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Die Abstimmung ist geschlossen. 35 υπέρ, 31 κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180. Σε δύο τμήματα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Thank you. Die Abstimmung ist geschlossen. 28 υπέρ, 38 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Η Abstimmung ist... 35 υπέρ, 31 κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Α, της ΔΕΒΕ, ναι. ΔΕΒΕ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. της ψηφορίας. 35 υπέρ, 31 κατά εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι σοσιαλιστές δεν συμμετείχαν. Ούτε ένας δεν ψήφισε. Σας παρακαλώ, σοσιαλιστές, ε, συμμετείχετε στην ψηφοφορία. 178 υπέρ. Ψηφίσατε όλοι, λέει ο Πρόεδρος. Πέρασε. 34 υπέρ, 30 κατά έγκρινεται. 179 υπέρ. Κατά. Άποχες ΔΕΒΕ DV11. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Άποχες. Α. Έλεγχος. Έλεγχος την 183. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 215. Πού είναι η 215. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος για την 215. Πέρας. 35 υπέρ, 30 κατά, εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αν ναι, δεν ψηφίζουν οι σοσιαλιστές, πολύ απλά δεν θα μετράνε οι ψήφοι του. Σας παρακαλώ, μας ε, κοστίζετε σε χρόνο. Μας καθυστερείτε. Σποραδικά συμμετέχουν κάποιοι σοσιαλιστές και αυτό μας καθυστερεί κάθε φορά. Σας παρακαλώ ζωμάδα να ψηφίζετε. Την 217 ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έλεγχος την 217. Πέρασε. 27 υπέρ, 37 κατά, Απορρίπτεται. Η 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 211. Πέρας. 32 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Άποχες. 214 υπέρ. Α, συγγνώμη, 212. Η 212 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρας. 35 υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 220 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Α, 21, 21. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. 23, γιατί το 23 θέλετε έλεγχο. Έλεγχο στην 23. Ποιο φώναξε ότι θέλει έλεγχο. Πείτε μου ποιο ήταν. Να σηκώνεστε και όρθιο, μιλάει ο κύριο Πάσκο. Ε? Incredible. 24. Ah, λοιπόν. 61 υπέρ, 4 κατά. Οριακό το αποτέλεσμα. 25 ε, υπέρ. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά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 Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3-1. Υπέρ. Κατά. Δεν ε, καταπίπτει. 31. Ε, Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 32. Ε, Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1. ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Πέρα ψηφοφορία 49 υπέρ, 11 κατά, μία παρατήρηση να κάνω, κοιτώντα την κατάσταση και σε άλλε επιτροπέ. Πρέπει να σα πω ότι εδώ πάντα είναι αρκετά γενναιόδορε οι πλειοψηφίε ε, για την υποστήριξη όλων των εκθέσεων και νομίζω ότι είναι θετικό σημάδι. Αυτό είναι σημάδι ε, συνεργασία συνεργασία μεταξύ του εισηγητή και των σκιωδών και των συντονιστών και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια καλή στάση. Γιατί έτσι κατά κανόνα μπορούμε να υποστηρίζουμε τις θέσεις μας ε, στο Κοινοβούλιο με ευρία πλειοψηφία. Και περνάμε λοιπόν τώρα στην ε, αναθεώρηση του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνο και για τον προπολογισμό. Η αρμόδια συγγήτρια από πλευρά μα είναι η Νίνα Τζιλ και θα σα παρακαλούσα να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Στο παρόν πλαίσιο και με τη σημασία που έχει η εξωτερική πολιτική αντιμετώπιση των πολλών κρίσεων που αντιμετωπίζονται, είναι σημαντικό η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να στείλει μία γνωμοδότηση συνεπή για το περιφές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήδη συναντήθηκα με τους Κιώδης, έγινε πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Πριν υποβληθεί το κείμενο σε 7 Απριλίου, συναντήθηκα και με πολλές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικές υπηρεσίες. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως σε κάποια από τα βασικά σημεία. Στο κεφάλαιο 4 καλύπτεται εξωτερική δράση. Πρόεδρε. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε λίγο, να ακούσετε αυτά που λέω. Καλό θα ήταν αυτό. Θα συνεχίσετε κουβέντα. Α, εντάξει. Είναι για τα χρήματα και έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, κεφάλαιο 4, εξωτερική δράση, τίτλος 4. Εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες κρίσεις και τις μεγαλύτερες ανάγκες. Και θα έλεγα η γειτονιά μας αντιμετωπίζει τεράστια αριθμό προβλημάτων. Φωτιά έχει αρπάξει, θα λέει η προβλήματα στην Ουκρανία, Συρία, Λιβύη, που δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα τα προβλήματα, ούτε και οι συνέπειες της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης. Τους τελευταίους μήνες, από όταν δημιουργήθηκε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε και μια αύξηση των φυσικών καταστροφών και όλοι αυτοί οι τομείς καλύπτονται στο κεφάλαιο 4. Να θυμηθούμε ποιες είναι οι πολιτικές μας προτεραιότητες. Αυτέ ψηφίσαμε στου προπολογισμού. Περιστρεφόταν γύρω από τι αναπτυξιακέ πολιτικέ. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λοιπόν την Αφρική και τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ταυτόχρονα, Έχουμε περικόψει άλλε πολιτικέ, Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση και την κρίση των προσφύγων. Θα πρέπει τα μακροπρόθεσμα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Εμεί, σαν Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αναλάβει υποχρεώσει να επιτύχουμε τους στόχους, τους στρατηγικούς. Ζητώ λοιπόν στο κείμενο να γίνει αναθεώρηση πραγματική του κεφαλαίου 4 Πρέπει να αυξηθούν τα ανώτατα όρια και των πληρωμών και των υποχρεώσεων. Τι το τρόπος μπορούμε να πετύχουμε τις ε, πολιτικές, πολιτικούς στόχους. Υπογραμμίζω και την ανάγκη να εξασφαλίσουμε και το εξή. Ότι οι απαντήσεις σε ανθρωπιστικά προβλήματα θα κινούνται εκ παραλίλου με την αναπτυξιακή διαδικασία. Ε, έχουμε απαιτήσει έναντι του κοινοτικού προπολογισμού λόγω των κρίσεων. Έτσι είδαμε ότι οι μηχανισμοί ευελιξίας οι παρόντες δεν αρκούν. Δεν αρκούν ούτε από πλευρά όγκου, ούτε όσον αφορά την ευελιξία για να δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις. Το μέσο της ευελιξίας έχει τελικά εξαντληθεί μετά από δύο χρόνια και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το διαπιστώσουμε. Πώς κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημιούργησε πολλά μέσα ad hoc, κατά περίπτωση δημιουργήθηκε και καταπίστευμα για τη Συρία, για την Αφρική και την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ένα για το μέσο για τους πρόσφυγες για την Τουρκία. Καταρχήν δεν έχω πρόβλημα με το καταπίστευμα. Ποια είναι η ανησυχία μου όμως αφήνει εκτός το κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα και θέλω να δω μηχανισμούς βάσει των οποίων μπορεί να επηρεάσει τα τεκτενόμενα το κοινοβούλιο και ίσως και να έχει θέση στα διοικητικά συμβούλια. Είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια. Λοιπόν, βασικά τι πιστεύω. Πιστεύω ότι στην αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να προτείνουμε ουσιαστική μεταρρύθμιση του μέσου ευελιξίας και του σχετικού μηχανισμού και να έχουμε ένα μόνιμο σύστημα που θα επιτρέπει την κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων όταν αυτοί απαιτούνται. Θεωρώ επίσης ότι η κατεπίγουσα χρηματοδότηση σε ανταπόκριση κρίση και για πρόβλεπτε καταστάσεις όλα αυτά πρέπει να καλύπτονται από ένα ειδικό εργαλείο που θα είναι εκτός των ανωτάτων ορίων του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αναφέρθηκα ρητά και στο εξής πρέπει να μπορούν να μεταφέρονται πόροι μεταξύ κεφαλαίων και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταποκρινόμεθα σε εξελισσόμενες κρίσεις. Κάτι που δεν είναι εφικτόν επί του παρόντος. Δοθέντως ότι έχουμε την διάμεση αναθεώρηση του εξωτερικού μέσου χρηματοδοτήσεως, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξετάσουμε και τις ανάγκες για καλύτερο συντονισμό, συνοχή, Και ποια θα είναι η μελλοντική αναθεωρητική διαδικασία. Χρειάζεται κάτι συντονισμό με άλλα λόγια. Μετά τι συναντήσει που είχαμε του Κιώδη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά ήταν τα βασικά θέματα που ετέθησαν. Έπρεπε να περιοριστούμε στο τι μπορεί να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Άρα έπρεπε να είμαστε πολύ συνοπτικοί και περιεκτικοί. Υπάρχει όμως δυνατότητα για τροπολογίες. Γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι θα υποβάλουν τροπολογίες και προσβλέπω στην αντίδραση και των άλλων συναδέλφων. Τι θεωρούν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Μπροκ. Εκτό μικροφώνου. Νομίζω ότι ω Επιτροπή Εκτορικών Υποθέσεων θα πρέπει να έχουμε μια μεγάλη και βρία βάση σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, γιατί κατά την αρχική κατάρτιση του σχεδίου 2014 και 2020 είχαμε κάποιες, ε, ε, δώσαμε κάποιες κατευθύνσεις ε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Και έγιναν περικοπές σε κάποιους τομείς όμως της εξωτερικής πολιτικής. Και σήμερα λοιπόν χρηματοδοτούμε ε, κάποια πράγματα από τα για των επόμενων ε, ετών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει με κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δούμε τι θα γίνει με το, το κεφάλαιο 4 και να δούμε και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και την ευελιξία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις διεθνείς μας ε, υποχρεώσεις δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων, τα τελευταία χρόνια. Και σε ό,τι αφορά ε, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της ε, προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, σε ό,τι αφορά την γειτονιά μας προς την Ανατολή και προς τον Νότο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε την εισηγήτρια και να θέσουμε τα ερωτήματα αυτά με σαφήνεια. Το λόγο λοιπόν έχει τώρα ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Αρνόντα Ντανζόν είναι ο σκιώδης ηγητής της ομάδας μας. Δυστυχώς κολλείται όμως σήμερα και μου ζήτησε να σας παρουσιάσω εγώ τις απόψεις του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Νίνα Γκίλ για το έργο της. Ο κύριος Τανζάν θεωρεί ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου έχει μεγάλη σημασία για να προσαρμόσουμε τις δημοσιονομικές μας προτεραιότητες ε, στις ανάγκες και με αυτή την αναθεώρηση θα δούμε τι μέτρα χρειαζόμαστε εκτάκτως να λάβουμε κατά προτεραιότητα και επίσης ε, ο κύριο Τανζάν στηρίζει ε, τις απόψεις κυρίας Γκίλ στα ακόλουθα σημεία. Την ανάγκη να αναθεωρήσουμε το ανώτατο όριο του τομέα 4. Ο προπολογισμό δεν μας επιτρέπει να ανταπεξέλθουμε στις δεσμεύσεις μας. Επίσης, το θέμα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι βέβαια προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να ε, χρηματοδοτεί εις βάρος άλλων θεμάτων. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και το μέσο ευελιξίας, ε, αποκαθιστώντας τη διαφάνεια. Επίσης, άλλο σημαντικό θέμα είναι για την ομάδα μας, είναι ο προπολογισμό που θα στηρίζεται στις επιδόσεις και ε, πραγματική διπόρη. Βλέπετε, μπερδεύει αγγλικά και γαλλικά ο κύριος Ταζό. Αυτό βέβαια θα απασχολήσει ιδιαίτερα την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ο κύριος Νταζό είναι ικανοποιημένο από το σχέδιο της κυρίας ε, Νίνα Γκίλ και θα επιμείνει σε δύο σημεία το, την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη μιας πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πλιανκοβίτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών να υποβάλω κάποιες παρατηρήσεις για την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Γκίλ. Καταρχήν, ε, είναι σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει στην ε, ανάγκη αναθεώρηση, διάμεση αναθεώρησης ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι τα τέλη του 2016 γιατί όταν αποφασίσαμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ούτε την σημερινή οικονομική κατάσταση ούτε μια σειρά παγκόσμιων κρίσεων που επηρεάζει την εξωτερική μας πολιτική και ασκεί νέες πιέσεις στον επταετή μας αυτό προϋπολογισμό. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το ισχύον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ε, χαμηλότερο από το προηγούμενο, το 2007-2013 και πρέπει το νέο πλαίσιο να προσαρμοστεί στις ε, νέες ανάγκες, στις νέες προκλήσεις και να εξασφαλίσει κάποια συνέπεια των, των πολιτικών μας με τις προτεραιότητες και τις αρχές μας. Ε, φαντάζομαι ότι η Επιτροπή θα ε, επικεντρωθεί σε μερικά μέτρα, θα δώσει έμφαση σε επενδύσεις και στην ανάκαμψη ε, και φυσικά δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην, ε, στον προβληματισμό για τον ε, προϋπολογισμό, αλλά να λάβουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε επίσης ε, το δυναμικό και την ικανότητα επιμέρους μηχανισμών των, του πολίτης δημοσιονομικού πλαισίου που ε, έχουν εξαντληθεί ιδιαίτερα στους τομείς 3 ε, και 4 εξαιτία της απρόβλεπτης μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Επίσης, ε, έχει περιοριστεί το περιθώριο λιγμών στα εσωτερικά όρια. Και μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποιες αυτοσχέδιες και πολύ ευρηματικές προτάσεις. Θα πρέπει όμως να διαφυλάξουμε την αρχή της ενότητας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Έχουμε μερικά trust fund εκτός του προϋπολογισμού για τη Συρία, την Αφρική και την πρόσφατη πρωτοβουλία για τη βοήθεια στην Τουρκία. Συμφωνώ με τις προτάσεις του κυρίου Πρέντα και του σκιώδου συζητητού μας, του κυρίου Ντανσάν, ότι χρειαζόμαστε ευελιξία και δυνατότητα άμεσης άσης προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις κρίσεις που τα τελευταία δύο χρόνια μας έδειξαν ότι πρέπει να επιταχύνουμε το ρυθμό αντίδρασή μας και να προσαρμόσουμε τα κονδύλια που έχουμε στον προϋπολογισμό στις ανάγκες μας. Γι' αυτό και είναι σημαντική η αναθεώρηση. Πάντως είμαι υπέρ του στενού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρότεινε και η συγκεκριά μας. Και ακριβώς επειδή έχουμε νέα παγκόσμια στρατηγική και στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, αυτό το θέμα θα αποτελέσει μεγάλη και σημαντική προτεραιότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο ρόλο μας ως σημαντικού ε, εταίρου στην παγκόσμια σκηνή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πλένκοβιτς. Η κυρία Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. ότι είχαμε υποστεί περικοπές αυτό που πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την κατηγορία 4 και έχουμε πολύ μεγαλύτερες απαιτήσει και ανάγκες. Το μήνυμα που έλαβα είναι ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικότεροι, να θέσουμε προτεραιότητες. Αλλά χρειαζόμαστε και αύξηση είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και να τα αποκρινόμεθα στις υποχρεώσεις, κυρίως όσον αφορά τα αναπτυξιακά και τους στόχους μας, που είναι τόσο σημαντικοί για μας, με αυτούς τους πόρους. Άκουσε αυτά που είπε ο κ. Πρέντα για την κατάτηση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων. Αυτά είναι θέματα που η Επιτροπή Προπολογισμών εξετάζει. Νομίζω ότι τα ζητήματα ασφαλείας πρέπει να λυθούν. Δεν πρέπει να ασφαλίσουμε μόνο τη γειτονιά μας, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό, αλλά να δούμε τι γίνεται και παραπέρα. Ποιο πρόβλημα έχουμε. Ότι τα μέσα δεν μας δίδουν αρκετά περιθώρια για ελιγμούς, είτε μεταξύ κεφαλαίων και κατηγοριών, είτε προσπαθώντας να εντοπίσουμε νέα μέσα και εργαλεία. Είναι σημαντικό κατά την άποψή μου να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι φάνταστη, να βρει λύσεις, να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στα διάφορα προβλήματα. Και εκεί που έχουμε οικονομικούς περιορισμούς και απαιτούνται περισσότεροι πόροι να βρεθεί λύση. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βρούμε περισσότερους πόρους για την κατηγορία 4 στα πλαίσια της αναθεωρήσεως. Διαφορετικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσουμε εμείς και να ανταποκρινόμεθα στις νέες κρίσεις. Ήδη προσθέσαμε και φυσικές καταστροφές που συνέβησαν. Από όταν ξεκίνησα την αναθεώρηση του κειμένου συνέβησαν και άλλα. Άρα πρέπει να ανταποκριθούμε και στις καινούργιες αυτού του είδους προκλήσεις που σας προανέφερα. Να καλύψουμε και αυτές. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνω να αλλάξουμε τις ημερομηνίε. προθεσμή υποβολής τροπολογιών. Πιο πριν. Και ψηφοφορία και, και αυτή μια εβδομάδα νωρίτερα. Βλέποντας τις διαδικασίες της Επιτροπής Προπολογισμών, αξίζει να είμαστε ε, πιο έγκαιρα έτοιμοι εμείς. Να μπορούμε να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα. Γι' αυτό, γιατί όχι. Κάντε το. Εδώ πολιτική διαμορφώνουμε, δεν κάνουμε διοικητική δουλειά. Η πρόκληση είναι η μετάφραση και η διερμηνία. Δεν το δέχομαι αυτό στην πολιτική, λέει ο κ. Μπροκ. Πάντα παρεμβαίνουν τέσσερις εβδομάδες. 19 Απριλίου είμαστε. Μπορούμε να έχουμε την ημερομηνία υποβολής τροπολογιών λίγες μέρες νωρίτερα. Τη μετακινήσουμε. Έτσι. Να επιταχύνουμε και τις διαδικασίες. Έχουμε γνωμοδότηση, όχι έκθεση. Και τι έχουμε τα 23 Μαΐου. Να ψηφίσουμε στη συνεδρία Επιτροπής στις 23 Μαΐου. Και έτσι η συγγήτριά μας θα έχει τη δυνατότητα τρεις εβδομάδες στη διάθεσή της μεταξύ αυτής της ημερομηνία για διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ωραία. Η ε, κυρία Γκίλ μου είπε η γραμματεία ότι θα είναι δυσχερέστατο να αλλάξουμε τις ημερομηνίες. Εγώ λέω ο ως Μπρόκ πιστεύω ότι η γραμματεία θα τα καταφέρει. Η ε, κυρία Γκίλ κοιτάξτε, αυτό αφορά και τους συναδέλφους. Αν ψηφίσουμε όταν δεν έχουμε έτοιμα όλα τα κείμενα σε όλες γλώσσες μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Θέλω να το σκεφτείτε, Πρόεδρε. Δεν θέλω η γνωμοδότησή μου να αψηφιστεί, να καταψηφιστεί, διότι κάποιος θα την αμφισβητήσει λέγοντας δεν έχουμε τη διερμηνία και τη μετάφραση και δεν ψηφίζω. Καμιά φορά πρέπει να κινούμεθα πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να σταματάει η γραφειοκρατία, Ρέκος Μπρόκ. Έχουμε από τώρα μέχρι 23 Μαΐου στη διάθεσή μας πάνω από τέσσερις εβδομάδες. Θα έπρεπε αυτό να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Δεν χρειαζόμαστε. Από τώρα με, παραπάνω, από τώρα μέχρι τις 23 έχουμε εβδομάδες. Ρωτήστε όλους τους κοιόδης των διαφόρων ομάδων αν οι διάφορες ομάδες συμφωνούν με αυτό, λέει η κυρία Εγώ ακολουθώ αυτό που μου είπε η διοίκηση. Και είπαμε, λέει Μπρόκ, ο να ζητήσουμε από τη διοίκηση να κινηθεί γρήγορα. Να ρωτήσω του Κιώδη. Δεν είμαστε θύματα τη διοίκηση, λέει και ο Κυρία Γκίλη, έπρεπε να ρωτήσω του Κιώδη. Διότι μπορεί να έχουν αντιρρήσει. Κύριε Σπρέντα. Είμαστε υπέρ της πρότασης ε, του Προέδρου. We have talked to the Secretary General who else θα το προσπαθήσουμε με τι άλλο. Αν δεν είναι δυνατόν θα το κάνουμε, αλλά μη τι άλλο το επιχειρήσουμε, ας το προσπαθήσουμε, κύριο Χόουιτ. Εγώ θα πρότεινα. Ε, έχουμε μια συνεδρία το πρωί. Γιατί δεν συνεννοείται η συντάκτη της γνωμοδότησης με τη γραμματεία και τους κοιόδης ηγητές και να μας το ανακοινώσει προς το τέλος της συνεδρίασης γιατί είναι θέμα πολιτικής, αλλά υπάρχουν θέματα, θέματα τακτικής. Καλύτερα να καταλήξουμε σε συμφωνία, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Έχουμε χρόνο σήμερα το πρωί, ας τα κανονίσει η συγγήτρια με τη γραμματεία και τους σκιώδει συγγητέ. To... Δεν θέλουμε. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα ε, να ε, επιταχύνουμε κάπως τα πράγματα, να πιέσουμε λίγο τη γραμματεία να βιαστεί. Ε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι για μια σύντομη γνωμοδότηση χρειαζόμαστε τέσσερι εβδομάδες για την ε, μετάφραση. Δεν το δέχομαι αυτό. Θα πρέπει να πιέσουμε την ε, διοίκηση, τη γραμματεία να φροντίσει και να είναι έτοιμη. Να το επιδιώξουμε. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό τη αναθεώρηση του προπολογισμού του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι από τα πιο σημαντικά θέματα, από τις πιο σημαντικέ ψηφοφορίε που θα κάνουμε πριν το καλοκαίρι. Γιατί θα επηρεάσει τα υπόλοιπα 2,5-3 χρόνια τη εξωτερική μα πολιτική. Και δεν είναι τυχαία γνωμοδότηση η έκθεση, παρά είναι σημαντική. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χρόνο. Το πιο σημαντικό είναι να διαμορφώσουμε τη γνωμοδότηση αρκετά νωρί, ώστε να μπούμε σε πρώιμη φάση των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή Προπολογισμού και αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε. Θα το τσεκάρουμε το πρωί με τη γραμματεία, με την ε, συντάκτρια. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά εγώ θα σας το δώσω. Η κυρία Γκίλ. Δεν έχω πρόβλημα με την αλλαγή της ε, ημερομηνίας και τις προθεσμίες, αρκεί να συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Προς το παρόν δεν βλέπω κανένα άλλο σκιώδη ηγητή. Μόνο το ΕΛΚ βλέπω εδώ. Μόνο το ΕΛΚ ε, τάχθηκε υπέρ της πρότασης. Οι υπόλοιποι σκιώδη ηγητές δεν αποφάνθηκαν. Ναι, είπαμε ναι. Και το χρονοδιάγραμμα δεν το αποφασίζουν οι σκιώδη συγγητές ούτως ή άλλως, αλλά η Επιτροπή. Ε, διαφωνώ. Είπα ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλες τις πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή. Και νομίζω ότι θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο ευγενείς απέναντι στους συναδέλφου σας, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε κάποια τα πράγματα. Το πρόβλημα, κυρία Γκίλ, είναι ότι έχει νόημα να επιταχύνουμε, να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τα πράγματα. Αν είναι εφικτό θα το καταφέρουμε. Αν δεν είναι θα τα αφήσουμε. Αλλά για πολιτικούς λόγους είναι σωστή επιτάχυνση. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα, λέει κυρία Γκίλ. Να μην έχουμε πρόβλημα όμως στη στιγμή της ψηφοφορίας. Καλώς, αργότερα θα δούμε την ε, διαδικασία. Η κυρία Βαλέρο. Δεν είμαι σκιώδης ε, εισηγήτρια των Πρασίνων. Αλλά περιμένουμε τη μελέτη για τη χρηματοπιστωτικά μέσα και τους μηχανισμούς η οποία αναμένεται για το Μάιο. Δεν θα ήταν σκόπιμο να δούμε και τα απορίσματα αυτής της μελέτης. Άλλο θέμα αυτό. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Μπίτι να ετοιμάσει στο δυνατό γρηγορότερα τη δική του έκθεση για αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα και τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς. Γιατί και ως προς αυτό το θέμα υπάρχει μια δυσφορία και δυσαρέσκεια. Πάμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 21, που είναι η συντάκτρια. Η κυρία Δεσαρνές είναι παρούσα. Έχετε το λόγο κυρία Σαρνές. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το θέμα είναι σημαντικότατο της ενισχύσεως των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα του Σέγγεν. Εδώ αγγίζουμε αυτό που είπατε προηγουμένως. Αποφασίστηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και έχουμε επιληφθεί αυτού και γι' αυτό προτείνω την ε, τοποθέτηση, την γνωμοδότηση αυτή, αναθεώρηση του καθεστώτος της διελεύσεως των συνόρων. Ο κώδικας Σέγκεν ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο. Η τροποποίηση θα επιτρέψει να έχουμε ενδελεχείς ελέγχου στα σύνορα ατόμων και στοιχείων μέσω φακέλων, αρχείων και βάσεων δεδομένων, των σχετικών βάσεων δεδομένων, αυτό θα αφορά τους υπηκόους Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τρίτων χωρών. Κατά βάθος μπορούμε να διερωτηθούμε όταν μιλάμε για αυτό σήμερα, γιατί αυτό δεν έγινε πριν. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή μεταρρύθμιση που είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλει ουσιαστικά να διατηρήσει το Σέγγεν, να ξαναδώσει μια αξιοπιστία στο Σέγγεν και την ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει προφανώς να έχει αποτελεσματικούς ελέγχους στα σύνορα ατόμων και δεδομένων. Λοιπόν, η γνωμότητα που προτείνω σήμερα ονόμα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έχει συμπεριλαμβάνει έξι τροπολογίε των φατήμων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σα να συντάξω τις τροπολογίες σεβόμενοι τι δικέ μας αρμοδιότητες και μετά συμφωνήσω αστικά με τι τρομολογηθήσει συζητήσει για να έχουμε μια έγκριση του κειμένου και κυρίω μια θέση σε ισχύ τάχιστη ε, της εν λόγω νομοθεσίας. Πάνω απ' όλα, συνολικά προτείνω έξι τροπολογίες, δύο τροπολογίες ε, για θεωρήσεις που πρέπει να προστατεύουμε βέβαια ε, τα δικαιώματα των παιδιών. Η τροπολογία 3 επενθυμίζει αιτιολογικέ αναφορέ. Θέλουμε να προστατεύσουμε όλου του Ευρωπαίου, είτε είναι υπήκο ενό κράτου μέλου τη Σέγγεν, είτε όχι, διότι η τρομοκρατική απειλή δεν περιορίζεται σε ένα μόνο κράτο μέλο και δεν απορρέει μόνο από εξωτερικού παράγοντε. Η τροπολογία 4 αφορά την αυτόματη επαεξακρίβωση τη διαταυτότητα των υπηκών τρίτων χωρών και την έξοδο αυτών. Αυτό είναι σαφέ το κείμενο. Οι τροπολογίε 5 και 6 αφορούν τις εξαιρέσεις όσον αφορά την αυτόματη εφαρμογή των μέτρων. Αναφέρεται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση που αυτή η διαβούλευση ε, συστηματική ε, ανάλυση των στοιχείων επηρεάζει τις ροές. Μπορούμε να προβλέπουμε παρεκκλήσεις. Η τροπολογία που προτείνω λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να παραμείνει μια εξαίρεση και να μην αποτελεί κανόνα και θα πρέπει η αξιολόγηση του κινδύνου να μπορεί να δικαιολογεί την εξαίρεση. Ιδού εν ολίγης, κύριε Πρόεδρε, αυτό που περιέχει αυτή η μεταρρύθμιση, προφανώς αυτό θα πρέπει να ειδωθεί σαν ένα σύνολο, όλα, όλα τα μεγάλα μορφώματα, όλα μεγάλα κράτη, ε, μορφώματα του κόσμου έχουν έλεγχο εξωτερικά σύνορα και θα πρέπει να περικοδοτηθεί από αυτό το μέσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόζει αυτό το μέτρο Προφανώς αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πεδίο ευρύτερο αποφάσεων πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση στο βαθμό του καλύτερο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να προστατευτούν οι πολίτες μας. Είναι απόφαση αυτή για το PNR που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε όλα αυτά τα κείμενα που καταφθάνουν κυρίως περί εναρμονωρήσεως ε, της προσπάθειας καταπολέμησης τρομοκρατίας και αρχεία για τους ξένους μαχητές, συνεργασία Eurojust ε, και Europol εντάσσονται στις πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά και πιστεύω ότι αυτή η μεταρρύθμιση κατά την άποψή μου του Σέγγεν καθυστέρησε ήδη να τεθεί σε ισχύ, να εφαρμοστεί και γι' αυτό ελπίζω ότι η δική μα Επιτροπή θα υποστηρίξει την όλη πολιτική βούληση για αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεσσαρνέζ. Ξεκινάμε με τι ομάδε. Ο κύριο Ντανζάν δεν είναι εδώ. Ο κύριο Πρέντα λοιπόν, ο συντονιστή μα θα παρουσιάσει τι θέσει του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Ενό Ντανζόν θα ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Ντεσαρνέ, τη συντάκτηρα τη γνωμοδότησης, για το έργο τη και να εκφράσει την αμέριστη υποστήριξη στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στόχο έχει την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, διατηρήσει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Θα πρέπει να βελτιωθεί ο μηχανισμό του Σέγγεν, ενισχύοντα τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, συστηματοποιώντα του ελέγχου στα σύνορα, ακόμη και για του υπηκόου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίε ε, του Σέγγεν δεν ε, εγγυώνται μόνο την ελεύθερη διακίνηση των ε, προσώπων, αλλά προβλέπουν και ενισχυμένου ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Αρνές ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό ο κύριος Νταζόν θα ήθελα να συνεργαστεί μαζί τη για να βαθύνει σε τρία κυρίως σημεία. Καταρχήν, συστηματική εξακρίβωση των στοιχείων από τα κρατημέλη των επικών κατά την έξοδο, όχι μόνο κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις κατάλληλες βάσεις ε, δεδομένων. Επίσης, συστηματική εξακρίβωση των στοιχείων των τρίτων, ε, ε, επικών τρίτων χωρών κατά την έξοδο, ώστε να μην αποτελούν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Και τρίτον, στοχευμένη εξακρίβωση στοιχείων των πολιτών, που είναι μια εξαίρεση ε, προκειμένου να μην διαταραχθεί απρόσκοπτη διακίνηση των προσώπων στα σύνορα. Ε, βέβαια, το θέμα της βάσης των δεδομένων είναι ε, πολύ δεσμευτικό. Πάντως, πιστεύω ότι και ελπίζω, κύριο Δαζάν, θα καταλήξουμε συμφωνία με το Συμβούλιο ώστε το νέο κείμενο να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρέτα. Ο σκιώδης εισηγητής από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι ο κύριος Πίτσουλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αντρέη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντάκτρια την κυρία Τεσσαρνές για την γνωμοδότηση αλλά και για, τι τροπολογίε για τις τροπολογίες της με τις οποίες συμφωνώ. Μετά τις τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στη Γαλλία και στο Βέλγιο διαπιστώσαμε τις αδυναμίες και τα κενά που έχει το σύστημα ασφάλειας και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα τη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών και αυτό έχει κενά και δυναμίες. Θα πρέπει λοιπόν να περιλάβουμε στις βάσεις των δεδομένων και τα απολεσθέντα ή ε, κλεμμένα ε, έγγραφα και να ενισχύσουμε ε, την, τους ελέγχους ιδιαίτερα και κατά την έξοδο, ιδιαίτερα όταν συγκεκριμένα πρόσωπα αποτελούν απειλή της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτός ο ε, συνδυασμός συστηματικών ε, ελέγχων ε, γράφων και προσώπων με βάση τις οικείς βάσεις δεδομένων θα εξασφαλίσει συνέργειες που μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατές. Οπότε με σωστή συστηματική ε, με σωστό συστηματικό έλεγχο και στοχευμένου ελέγχους θα ενισχύσουμε την ασφάλεια. Βέβαια τέτοιες, τέτοιοι μηχανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτόματα αναφέρεται. Αυτό ίσως έχει κάποιες τεχνικές, τεχνολογικές και διοικητικές συνέπειες ό,τι αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ιδιαίτερα στις, ε, στα σημεία ε, διέλευσης που είναι ε, τα πιο πυκνά στη διακίνηση. Θα Βέβαια η ασύρμα τεχνολογία δεν επιτρέπει αρκετά ταχύτατη ε, εξακρίβωση των στοιχείων. Ε, χρειάζεται λοιπόν να βελτιώσουμε και αυτό το τεχνολογικό σημείο και ιδιαίτερα στις εποχιακές περιόδους εχμής ίσως οδηγήσει σε συμφόρηση του συστήματος. Βέβαια προηγουμένως είχαμε ελάχιστες, ε, ελάχιστους ελέγχους και πολύ σποραδικούς των ταξιδιωτικών αγράφων αλλά θεωρώ ότι η νέα πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τεκμηριωμένη και σωστή και θέλω αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ τον Ινώ. Η κυρία Βαλέρα τώρα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήμουν ικανοποιημένη αν θα μπορούσαμε να μαθήσουμε τους εσωτερικούς ε, ελέγχους ε, στα σύνορα μεταξύ Σουηδίας και Δανίας, ε, για παράδειγμα. Αλλά προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι εξωτερικοί έλεγχοι. Αυτό που πιστεύω ότι είναι σημαντικό στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε την ακυρεότητα των ανθρώπων. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις μορφές. Θεωρώ λοιπόν ότι η τροπολογίε που κατέθεσε ο εισηγητή κινούνται προ την κατεύθυνση αυτή και επ' αυτού θα επικεντρωθούμε. Πώ μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα ε, παραβιάζει τα δικαιώματα και την εγκαιρότητα των ανθρώπων. Ευχαριστώ κύριε Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι κατατεθήσει τροπολογίε γενικώ ε, κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση και υπό την έννοια αυτή πρέπει να υποστηριχτούν. Όμως Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτή η ενέργεια είναι το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να μην επιτρέπεται η αλεξέλεγκτη ροή όλων αυτών των λαθραμεταναστών και των ανθρώπων που θέλουν ουσιαστικά να εισβάλλουν στην Ευρώπη. Και αυτή η προσπάθεια, αυτή η αποτροπή της ε, αθρώας εισβολής αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών που έχουν τα εξωτερικά σύνορα. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δώσουμε πρώτη προσοχή και μετά όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Διότι βεβαίως κανείς δεν θέλει να παραβιάζει δικαιώματα, κανείς δεν θέλει να μην προστατεύει τα παιδιά, κανείς δεν θέλει να μην προστατεύει τις γυναίκες και κανείς δεν επιθυμεί να δημιουργήσει κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρώπων. Όμως πρέπει να εξομαλυνθεί πρώτα η κατάσταση και κατόπιν να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετήδια. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών για το θέμα αυτό και κύριε Αντεσόρνε, θα θέλετε να πάρετε το λόγο για να συμπληρώσετε. Ευχαριστώ, απλώς ε, διαπιστώνω με ικανοποίηση ε, και χαρά ότι κατά βάθο όλοι ε, πιστεύουμε το ίδιο πράγμα και υπάρχει μια συνοχή και σύμπνοια για αυτό το θεμελιώδη ζήτημα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν ε, θέλουμε να διαφυλάξουμε το χώρο του Σέγγεν θα πρέπει να έχουμε συστηματικούς και ευρυθείς ελέγχους στα σύνορα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι εκ των όνων προϋπόθεση για να διαφυλαχθεί η ελευθερία διακίνησης. Χρειαζόμαστε πραγματικούς αποτελεσματικούς ελέγχους στα σύνορα και των προσώπων και των στοιχείων των δεδομένων και χαίρομαι για την συνένεση που διαπίστωσα και ευχαριστώ τους και οδησηγητές ε, που έλαβαν το λόγο. Ένα άλλο θέμα είναι το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής ή ε, η πολιτική ασύλου της Ευρώπης, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Θερμά ευχαριστώ σε όλους γιατί βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους πολίτες και για την λειτουργία των εξωτερικών συνόρων και προφανώς για τη λειτουργία του συστήματος Σέγγεν. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι στα πλαίσια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, θα λάβουν υπόψη όλες τις διαφορετικές αυτές απόψεις και αυτό που θα προκύψει ως αποτέλεσμα από την Επιτροπή Εξωτερικών ε, Υποθέσεων να θυμόμαστε ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την ε, ε, ε έκθεση αυτή είναι 28 Απριλίου και προβλέπεται στις 24, η προβλέπεται στις 24 Μαΐου προς το παρόν. Άρα έχουμε κάποια δεκαετία ημέρες για να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για την έκθεση της κυρίας Δεσσαρνέζα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε το 21 και με ενημερώνουν ότι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Αλλά ο κ. Βίγκαντ, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΤ, δεν είναι παρόν ακόμα και μέχρι τις 11 και 4 θα καταφτάσει. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, να, να επισημάνω τον σημαντικό αριθμό των μελών της Επιτροπής μας που είναι ακόμα παρόντες. Ναι, είμαστε καλύτεροι, αλλά είμαστε έξι μόλις στον αριθμό. Ναι, είναι μια διαπίστωση ε, για την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώ. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για καφέ. Τα λέμε στι 11 και 4 και πάλι. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε μία παρανόηση ως προς την ημερήσια διάταξη και κάποιοι συνάδελφοι αποχώρησαν. Ελπίζω ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. Κανονικά δεν έπρεπε καν να είχαν φύγει. Nichtsdestotrotz möchte Sie informieren, Herr Offiziell, θα ήθελα να σας ενημερώσω και επίσημα ότι ο κύριος Γιούνος είναι στον... Ε, είναι ε, οδεύει προς το Βερολίνο για ιατρική παρακολούθηση. Μετά από 1,5 έτος ε, μπορεί πλέον ε, να μεταβεί στο εξωτερικό για ιατρική παρακολούθηση. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί καλή εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της εργασίας που κάναμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Εξωτερική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τώρα έχει αναλάβει τα ιατρικά έξοδα μαζί με το Κοινοβούλιο προκειμένου και σε ένα τέτοιο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επιτευχθεί ένα εύλογο αποτέλεσμα, το θεμητό και ευχθέω να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα χωρί μεγάλε εισαγωγή να δώσω το λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Βίγκαντ. Äh, ähm, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ως ε, πρώην ε, δεν σύμβουλος σύμβουλο από την Ανατολική Γειτονία. Πρέπει να πω ότι με αγγίζουν ιδιαίτερα οι καλέ ειδήσει που μα αναφέρεται για τον κύριο Γιούνο και συνεργαστήκαμε επί μακρόν πολύ αποτελεσματικά για τέτοια ζητήματα και για άλλα ε, ε, περίπλοκα ζητήματα σε διαφορετικό Αζερβαϊτζάν. Τώρα όμω είμαι διευθύνοντα σύμβουλο για την Ασία και τον Ελληνικό. Θα μιλήσω για τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδίας ήταν η πρώτη σε δύο χρόνια που είχαμε σύνοδο κορυφής με την Ινδία μετά το 2012 και η πρόσκληση από την Επιτροπή σας αντικατοπτρίζει το μεγάλο ενδιαφέρον της Επιτροπής σας για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Και έχουμε πολλές δραστηριότητε του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις σχέσεις με την Ινδία. Αυτή η Σύνοδος Κορυφής έλαβε χώρα μία εβδομάδα μετά τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες στις 30 Μαρτίου και έδωσε πολιτική όθηση στις προσπάθειες και ήταν και ο βασικός σκοπός των δύο πλευρών. Γνωρίζουμε και δύο ότι αυτή η σχέση έχει σημασία. Ήταν επικοδομητική, θετική σύνοδος κορυφής, με πλούσια αποτελέσματα και εκφράστηκε πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές να αναπτυχθεί πλήρως η σχέση Πετύχαμε τα αποτελέσματα, πολλά αποτελέσματα, θα τα παριθμίσω, αλλά να υπογραμμίσω ότι είχαμε όχι μόνο τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρόεδρο μου, είχαμε και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την είπατε εκπρόσωπο την κυρία Μογκερίνη που συμμετείχαν από την δική πλευρά. Είχαμε τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας. Έχουμε δήλωση, κοινή δήλωση. Δείχνει ότι θέλουμε να αυξήσουμε τη συνεργασία. Και αυτό σε πολλούς τομείς. Θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τους νέους προσανατολισμούς που ακολουθεί η Ινδία, η νέα κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό Μούντι. Θέλουν να κάνουν αλλαγέ στην Ινδία σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, να εξυγχρονιστεί η χώρα. Και αυτό θα το συνδυάσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Να στηρίξουμε την καινοτομία και την ανάπτυξη θέλουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να συνδυάσουμε τις προσεγγίσεις. Εντοπίσαμε μελλοντικέ δράσεις Έχουμε κοινό πρόγραμμα δράσης μέχρι το 2020. Έχουμε συγκεκριμένο, και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Έτσι θα κινηθούμε την επόμενη πενταετία βάση των κατευθύνσεων. Τι θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Ότι θα κινηθούμε και οι δύο πλευρές, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε τις συγκεκριμένες δράσεις που αποφασίσαμε. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τρομοκρατία. Θέλουμε ο ένας να είναι στο πλευρό του άλλου στην προσπάθεια αυτή κατά πολεμήσεω τη τρομοκρατίας. Να υπενθυμίσω ότι σκοτώθηκε και ένας Ινδός υπήκοος της ε, πρόσφατες επιθέσεις. Υπεγράφει κοινό θεματολόγιο για την κινητικότητα και μετανάστευση. Είναι σημαντικό μήνυμα όσον αφορά την παγκόσμια μετανάστευση και την κρίση των προσφύγων. έχουμε εξαίρεση θεωρήσεων διαβατηρίων για διπλωματικά διαβατήρια και συζητήσαμε το θέμα επανεισδοχής υπηκών των δύο πλευρών. Έχουμε κοινή δήλωση για σύμπραξη για τα θέματα του ύδατος. Θέλουμε πιο πολύ εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν για τη διαχείριση των υδάτων στο δέλτα του Γάγκη και σε άλλους ποταμούς. Συμφωνήσαμε επί κοινής για καθαρή ενέργεια και για το κλίμα. Εκεί εστιαζόμαστε στη συνεργασία για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Προβλέπονται και συγκεκριμένες προσπάθειες στη χώρα για να κινηθεί η χώρα προς την χρήση ανανεωσίμων ε, πηγών ενέργεια και για να μειώσει τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρωπο, Ο πρόεδρο Χόιερ ήταν εκεί για να είναι μάρτυρας τη υπογραφή τη πρώτη δόσεω 450 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, για κάποιες επενδύσεις στην ειδική πόλη Λάκνορ. Θέλουμε ορατότητα μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα έχουμε μια νέα αντιπροσωπεία που θα ανοίξει στο Νέο Δελχή. Πολλοί παρατηρητέ θέλουν να βρούμε και κάποια λύση όσον αφορά τη συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο. Οι ηγέτε όμω δεν ήταν ακόμα σε θέση να προχωρήσουν εκεί παρά τι διαβουλεύσει πριν από τη Σύνοδο Κορυφή. Υπάρχει δέσμευση των ηγετών όμω να κινηθούν προ μια μελλοντική επανάληψη και προώθηση των διαπραγματεύσεων θα γίνει η προσπάθεια σε υπουργικό επίπεδο. Να δούμε που χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Και στη σύνοδο G20 στη Τζάνα το Σεπτέμβριο να γίνουν συζητήσεις στο περιθώριο και να προχωρήσουμε. Και οι δύο πλευρές διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευκαμψία για να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια για τις συζητήσεις. Συζητήσαμε εκτενώς την τρομοκρατία. Θεωρήσαμε ότι είναι παγκόσμια απειλή. Χρειάζεται συνεργασία διμερής και πολυμερής. Συζητήσαμε την πολιτική γειτονία, τη γειτονιά της Ινδίας, Αφγανιστάν, Πακιστάν και η διάσκεψη των Βρυξελών για το Αφγανιστάν είναι πολύ σημαντική. Συμβάλλει η Ινδία στις προσπάθειες. Συζητήθηκε και η Ουκρανία όμως. και θέματα που αφορούν την νότια γειτονιά μα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα συζητήσαμε, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα των φύλων, ε, μη διακριτική μεταχείριση και τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται. Χρειάζεται συνεργασία στα διεθνή φόρα. Θέλουμε πρακτική εφαρμογή όλων αυτών θα γίνει μια συνάντηση για θέματα ανθρω... ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα γίνουν και άλλοι διάλογοι με την Ινδία πάνω σε αυτό. Κάποια μέλη παρακολούθησαν την συζήτηση για τους α, ε, Ιταλούς πεζοναύτες. Αναφέρεται σχετικό στοιχείο στην κοινή δήλωση. χρειάζεται και οι δύο πλευρές να καταβάλουν προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος. Στην κοινή δήλωση αναφερόμαστε και στους Εστονούς και Βρετανούς ε, φύλακες ε, ασφαλείας. Στην περίπτωση των Ιταλών ε, πεζοναυτών θα πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία επιλύσεως των διαφορών και περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εκφράστηκε επιθυμία να προχωρήσουμε σε βάθηση των σχέσεων. Θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των επιχειρηματιών και των δύο πλευρών. Να εφαρμόσουμε ένα ευρύ θεματολόγιο. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου είναι κρισίμου σημασία. Θα δοθεί ιδιαίτερη πολιτική προσοχή με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και θα δοθεί και υποστήριξη από τα κοινοβούλια και των δύο πλευρών. Και ο πρόεδρος Σούλτς είπε ότι θα μεταβεί εκ νέου στην Ινδία. Καλωσορίζεται η στενότερη συνεργασία των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ινδίας. Κάτι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Το συμφωνήσαμε. Ο πρόεδρος Μούντι με τον Τούλτς συμφωνήσαμε από αυτού. Και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σχέση με την Ινδία ελπίζουμε να έχει και ομόλογη πλευρά στην Ινδία για να συνεχιστούν ε, οι συνομιλίες και να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει αυτή η ε, στατηγική εταιρική σχέση. Αυτά και ευχαριστώ. Εκτό μικροφώνου ο κύριος ε, Μπροκ. Η κυρία Γκίλη, μάλλον ο κύριος Βανόρντεν πρώτα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε τον κύριο Βίγκαντ για την ενημέρωση. Χαιρόμαστε για την διεξαγωγή αυτή τη ε, Συνόδου Κορυφή. Ήταν η πρώτη μετά από τέσσερα χρόνια. Και μάλιστα το ανακοινωθέν ήταν <laughs> μακροστελέστερο από τις, ε, ή τις συζητήσεις, γιατί ήταν σχετικά σύντομη η τι συζητησεις γιατι Κορυφής. η συνοδος κορυφη είχατε και ένα δείπνο εργασία, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί ήταν που ήρθε και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετείχε στην Αμυγυρή. Πριν την Σύνοδο Κορυφής είχαμε ευκαιρίες συνάντησης μεταξύ πολλών ευρωβουλευτών και βέλγων βουλευτών που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ιδέα παρουσία του Πρωθυπουργού Μόντε. Και περάσαμε τρία τέταρτα μαζί του συζητώντας ε, πριν την ε, Σύνοδο Κορυφής. Και στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό Μόντι, επισηρεμάναμε τις ανησυχίες μας ε, και επαναλάβαμε την ελπίδα μας να σημειωθεί πρόοδος στην ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Περιμένουμε ότι αυτό θα ήταν από τα σημαντικότερα θέματα της Συνόδου Κορυφής και μας απογοήτευσε το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε αισθητή πρόοδο στα θέματα αυτά. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μόντι εξέφρασε τη δέσμευσή του υπέρ της προόδου στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Ένας συνάδελφος μάλιστα προσπάθησε να προκαλέσει τον Πρωθυπουργό Μόντι αναφέροντας ε, τη θέση του, ε, ζητώντας τη γνώμη του για το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Μόντι απήχε και δεν έλαβε θέση. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, Μέχρι στιγμής είχαμε μία de facto αποτελμάτωση από το καλοκαίρι του 2013. Και ούτε το χρονοδιάγραμμα, αλλά ούτε και η ουσία της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών δεν αναφέρθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής. Βέβαια, καλή αναγνώριση για την ανάγκε μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερης αλλά χρειαζόμαστε ένα πραγματικό χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις, τις μελλοντικές δράσεις. Βέβαια, εκτοξεύονται ολοκατηγορίες ε, για την έλλειψη πρόοδου και από τις δύο πλευρές. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε κολλήσει και είναι απογοητευτικό που δεν σημειώθηκε πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, Βουλής της Ινδίας, εκεί είχαμε πρόοδο. Στείλαμε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία μας στην Ινδία και μάλιστα ε, εκφράσαμε την πρόσκληση του Προέδρου ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Πρόεδρο της ε, Ειδικής Βουλής, την Πρόεδρο, ήρθε και φαντάζομαι το Δεκέμβριο του 2016 θα ανταποδώσει την επίσκεψη ο Πρόεδρος Σούλτς. Από αυτή την άποψη υπήρξε πρόοδος στη σύσφυξη των σχέσεων με την Ειδική Βουλή. Γενικώ όμως είμαι απογοητευμένος κυρίως ε, εξαιτίας έλλειψη πρόοδου στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, που αποτελεί κεντρικό άξονα των ε, σχέσεών μας με την Ινδία. Και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα σημειώσουμε πρόοδο και στο θέμα των ελεύθερων συναλλαγών. Ευχαριστώ. Ήρθε η σειρά μου τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο Τζέφρι. Και σε ό,τι αφορά την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ελεύθερου Εμπορίου, κρίμα που δεν είχαμε πρόοδο. Πάντω το πιο θετικό είναι ότι μετά από τέσσερα χρόνια επιτέλου ε, έγινε μία σύνοδο κορυφή. και δόθηκαν κάποιε στρατηγικέ προοπτικές στη σχέση μα με την Ινδία. Και χαίρομαι ε, και την πρόταση για το σχέδιο δράσης, για την ενέργεια, το περιβάλλον, ε, τη συνεργασία, την τρομοκρατία. Ίσως χρειαζόμαστε πιο ευρύτερη, μακρόπνοη ε, πρόπτικη στρατηγικής, όχι επικεντρωμένη στα βραχυπρόθεσμα. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα η Ινδία θα υπερκεράσει από οικονομική άποψη την Κίνα. Οπότε καλό θα ήταν να επενδύσουμε στην προβολή των σχέσεών μας με τη χώρα αυτή. Και λυπούμε που και απογοητεύτηκα που δεν έγινε καν συνέντευξη τύπου δεν δόθηκε μετά την Σύνοδο Κορυφής. Κάτι ασυνήθιστο και αρκετά παράξενο. Και νομίζω ότι και για τις δύο πλευρές είναι σημαντικό να αναδείξουμε την αξία και τα προτερήματα αυτής της σχέσης. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δελχή. Ε, αλλά τα θεσμικά όργανα εκατέρωθεν ε, δεν προβάλλουν δεόντως αυτές τις σχέσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια γεωπολιτική συνειδητοποίηση της σημασίας που έχουν οι σχέσεις μας με την Ινδία. Καλά όσα γίνονται ε, και θετικό το άνοιγμα του γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μια και η Ινδία δεν είναι πια στο ερευνητικό πρόγραμμα δράσης, ε, στο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο το υπαριθμών 7. Καλό θα ήταν να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας εκεί. Μία από τις πρωτοβουλίες μας ε, για τη σύσταση του EPTC, ε, που τώρα θα κλείσει, ήταν κάτι που μας βοήθησε για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις εταιρείες γενικά να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και στην ειδική αγορά. Χάσαμε όμως μια ευκαιρία μια και δεν έγινε συμφωνία για την πέμπτη γενιά. Αντίστοιχη ε, αυτή που έχουμε με την Κίνα, Βραζιλία και Νότια Κορέα. Δεν έχουμε τέτοια συμφωνία πέμπτης γενιάς. Βέβαια, έχουμε επικάλυψη με το ψηφιακό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τεράστιο δυναμικό. Και στην συνάντηση που προανέφερε ο Τζέφρι, παρουσία του Ινδου Πρωθυπουργού, συζητήθηκε ε, κάπως το πεδίο εφαρμογή και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, μια και η Ινδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση ε, στον ψηφιακό τομέα και ε, ο τομέας αυτός είναι από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ινδίας. Καλό θα ήταν λοιπόν να τρέξουμε στα θέματα αυτά του ψηφιακού θεματολογίου. Φαντάζομαι έχετε ένα πρόγραμμα για τις επερχόμενες ε, συνόδους κορυφής. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί και πάλι μια τέτοια κοιλιά, ένα τέτοιο κενό τετραετίας Ελπίζω, αν μη τι άλλο, με αυτή τη Σύνοδο Κορυφή να θεσμοθετηθούν πιο τακτικέ σύνοδο Κορυφή, ώστε να διερευνήσουμε περαιτέρω του επιμέρου τομεί. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Θα Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα ακρηγορήσω, διότι προλαλήσαντες ε, ήδη είπαν αυτά που έπρεπε να υποθούν ανησύχησα κάπως από τη μικρή δυναμική των σχέσεων μας με την Ινδία. Δεν θα πω ότι έχω καθησυχάσει σε σχέση με το πρόβλημα αυτό. Χαίρομαι όμως παρόλα αυτά διότι είδα ότι επετεύχθη η πρόοδος. Υπάρχει, υπάρχουν δυνατότητες αυτή τη σχέση με την Ινδία, τεράστιες δυνατότητες υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε επίπεδο κρατών μελών που ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο όσον αφορά τις δυνατότητες συνεργασίας. Βλέπω ότι υπάρχει δυναμικό, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτό. Βλέπω επίσης το όλο θέμα στα πλαίσια της διασκέψεως των Παρισίων. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά για το πρασίνισμα, όπως αποκαλείται, της συνδικής οικονομίας και νομίζω ότι η Ινδία θα παίξει έναν πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων των Παρισίων. Είμαι πολύ ικανοποιημένο λοιπόν που βλέπω ότι έχει επιτευχθεί η πρόοδος και χαιρετίζω αυτές τις ειδήσει όσον αφορά το άνοιγμα του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τάπεζας Επενδύσεων στο Νέο Δελχή Είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι βλέπω ότι αυτή η συνεργασία ξεκινά και πιστεύω ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η δυναμική αυτή στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος, λέει ο κ. Μπροκ, εκτός μικροφώνου. Να ξεκινήσω κι εγώ. Ε, να δώσω το λόγο σε συνάδελφο που τον έχει ζητήσει, αλλά ε, δεν ε, είναι εδώ. Δεν θα θέλα. Θα θέλετε να απαντήσετε, κύριε Βίγκαντ. Η απάντηση σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρία Τζίλα νομίζω ότι αφορά και τα αφορά όλους ε, τους ευρωβουλευτές, γι' αυτό λοιπόν θα απαντήσω σε, στην ερώτησή τη. Καταρχά λοιπόν έχουμε και το θέμα τη απογοήτευση που εξέφερε ο κ. Φανόρντον. Και εμεί συμφωνούμε και είμαστε εξίσου απογοητευμένοι, γιατί θα θέλαμε οι διαπραγματεύσει για τη ζώνη ελευθερού εμπορίου να ε, ξαναξεκινήσουν με πλήρη ταχύτητα εννέα χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων και τρία χρόνια μετά από την τελμάτωσή τους Ίσως ε, είχαμε και τους ε, βασικούς διαπραγματευτές και τον επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης ε, Εμπορίου και την Ινδούς εμπειρογνώμονες για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Αλλά παρά το γεγονός αυτό υπάρχει πολιτική βούληση και έχουμε ξαναποκτήσει μια κάποια ταχύτητα και όντως η Ινδία θέλει να ανοίξει την αγορά της με πολύ προσεκτικό τρόπο και φοβάται ιδιαίτερα την γρήγορη απελευθέρωση. Είναι λοιπόν συνεκτική και συνολική η προσέγγιση μας σε ό,τι αφορά ε, την απελευθέρωση του εμπορίου και τη συμπερίληψη των επενδύσεων και αυτό έχει να κάνει με τις δομικές ε, αρχές του ζητήματος. Η, Ινδία θέλει περιορισμένη απελευθέρωση σε ό,τι αφορά την κλασική, το κλασικό πεδίο εφαρμογή ε, τη απελευθέρωση, τη ζώνη ελευθερίου εμπορίου. Εμεί είμαστε πιο γρήγορη, πιο ανοιχτή. Και θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Ένα βασικό ζήτημα είναι τα αυτοκίνητα, τα εξαρτήματα αυτοκινήτων από δική μας πλευράς ε, και θέλουμε ε, σημαντική πρόσβαση των παροχών μας στην αγορά εργασίας. Και αυτά είναι τα δύο βασικότερα ζητήματα. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλα, αλλά συνεχίζονται οι εργασίες σχετικά αισιόδοξο. Αν ε, αφιερώσουμε χρόνο και προσπάθεια, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά. Σε ό,τι αφορά και την σύνοδο των G20, να μπορέσουμε να στείλουμε τα σωστά μηνύματα για την ε, επιτάχυνση της διαδικασίας και την επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Για τους υπουργούς και τους βασικούς αξιωματούχους που προσπαθούν να βρουν τη σωστή μορφή συνεργασίας. Και φυσικά είναι τεράστιο το δυναμικό, έχετε δίκιο. Γιατί αναπτύσσεται γρήγορα η χώρα και οι ευκαιρίες της αγοράς είναι τεράστιες. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κυρίας Τζίλ τώρα. Η έλλειψη συνέντευξης τύπου όταν στο γεγονός ότι ήθελε η ειδική πλευρά να, γίνεται, να γίνει συνέντευξη τύπου χωρίς ρωτήσεις. Ήταν στενό το χρονοδιάγραμμα μεταξύ της διμερούς βελγικής ε, επίσκεψης των συναντήσεων με, τον, ε, με τους ε, εκεί και άλλες επισκέψεις, αλλά όλα αυτά δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε από αυτό και γι' αυτό δεν διοργανώθηκε συνέντευξη τύπου. Και η προβολή θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τις ενεργειές μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ινδία. Για την Ινδία θα πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, όχι μόνο συνέντευξη τύπου. Επίσης η κυρία Τζίλ αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό και Επιχειρηματικό Κέντρο. Το κέντρο αυτό δεν πρόκειται να κλείσει. Θα συμμετέχει ενεργά στην διαχείριση και εφαρμογή της διακήρυξης. Όπως σε κάθε έργο, φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από κάποιο διάστημα ελέγχει και τη βιωσιμότητα και την εφικτότητα του έργου για να συνεχίσει τη χρηματική υποστήριξη αλλά θα είναι αυτοσυντηρούμενο το κέντρο. Είμαστε βέβαιοι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη σημαντική έκθεση στην Ινδία, 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμμετοχή στο μετρό, 1,75 προβλέπεται και θα είναι αυξητική αυτή η τάση. Και τέλος χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Πέτερλε παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν ήταν απογοητευμένος για τη μία αξιοποίηση του δυναμικού μας, πλέον είναι ικανοποιημένο ότι έχουμε αναπτύξει μία σωστή ταχύτητα και ότι υπάρχει προθεμία συνεργασία και μάλιστα σε συνεκτικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, αυτή η σχέση, αλλά επιφυλάσσει πάρα πολλέ δυνατότητες και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και νομίζω ότι με την καινούργια ατζέντα έχουμε ένα βασικό πρόγραμμα εργασία το οποίο θα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε αυτό. Είναι μια δοκιμασία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις ικανότητες της ε, από την ειδική πλευρά κατά πόσο μπορούν να ξεπεράσουν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τις λοιπές δυσκολίες. Είμαστε λοιπόν δεσμευμένοι και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ελπίζω σε μισό χρόνο να μπορέσουμε να σας αναφέρουμε ότι θα έχουμε πετύχει θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος, δεν θέλει άλλος να μιλήσει. Συμφωνώ νομίζω με τους τρεις ομιλητές. Θα συμφωνείτε κι εσείς όπως είπατε πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη προτεραιότητα η Ινδία για μας, για λόγους πολιτικούς και οικονομικούς. Η Κίνα ακόμα δεν έχει γίνει δημοκρατική χώρα και δεν επικρατεί το κράτος δικαίου. Αυτό είναι ένα όφελος αντιθέτως που έχει ένα θετικό στοιχείο που έχει η Ινδία. Γι' αυτό πιστεύω μακροπρόθεσμα ότι η Ινδία έχει τις ίδιες δυνατότητες όπως και η Κίνα Τουλάχιστον αυτό. Και δεν θα πρέπει αυτό να το αγνοήσουμε και να μείνουμε πίσω. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να μας βοηθήσετε τόσο ώστε να το βάλουμε σαν σημείο προτεραιότητα στην ατζέντα μας, την Ινδία. Ευχαριστώ, ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Θα τα ξαναπούμε στις 3. Καλό μεσημέρι, καλή όρεξη.